Ευχαριστώ. Παρακαλώ να καθίσετε. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να καθίσετε κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας η γραπτή απάντηση στην ερώτηση 49 για το θέμα των ζώων που σφαγιάζονται έχουν υποβληθεί με την πλειοψηφία των υπογραφών των μελών των Ευρωβουλευτών και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό μεταδίδεται στους υπευθύνους και θεωρείται σαν το αποδεδειγμένο κείμενο. Ο κύριος Σλούτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια συνδυασμένη προσπάθεια του Νταν Τζόργκερσεν, την Έστε Ντελάλινγκε και του Ανδρέα Τζανόνι και του υποφαινομένου. Ε, ευχαριστώ όλου όσου το υπέγραψαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 8 χρόνια είχε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι όπου μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο μεταφορών θα πρέπει να δημιουργήσουμε την κατάλληλη πολιτική πίεση γι' αυτό. Το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και το Κοινοβούλιο ετοίμασε αυτέ τι υπογραφέ. Ε, πάνω από το μισό κοινοβούλιο και αρκετοί υπουργοί και επομένως ε, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πολιτική πίεση είναι προς εσάς. Σας παρακαλώ δώστε μας αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Αυτό ήταν ε, τώρα ο κύριος Γιώργενσεν. Ευχαριστώ. Δύο επίτροποι στάθηκαν εδώ στην Ολομέλεια και μας είπαν ότι θα υπάρξει πρόταση νομοθεσία στον τομέα αυτό. Ε, τη ζητήσαμε δύο φορές και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα ε, τόσα εκατομμύρια πολίτες ζητούν νέα νομοθεσία. Εμείς ε, στην Ολομέλεια έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε αυτή τη νομοθεσία. Δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η γραπτή, ε, η γραπτή ερώτηση 50 των Μοντάλτο Βέλτα ε, Τάκουλα ε, σχετικά με το πρόγραμμα